Καλησπέρα συνάδελφοι. Ξεκινάμε το σημείο 17 για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και τους μεθοριοφύλακες. Έχουμε τον αντιπρόεδρο τον κύριο Τίμερμανς, τον καλωσορίζουμε θερμά. Θα παραμείνει μαζί μας για τα αρχικά σημεία πριν φτάσουμε στο σημείο για την Ουγγαρία που θα μας μιλήσει. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Φραντς που είναι εδώ για την Ευρωπαϊκή Μεθοριοφυλακή και ακτοφυλακή Ρομπέρτα Ρομπέρτο Ματσόλα είναι η Ρομπέρτα Ματσόλα μάλλον και θα τη δώσω το λόγο για να μα ενημερώσει για τι διαπραγματεύσει στον τριμερή διάλογο. Λοιπόν, Ρομπέρτα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να καλωσορίσω τον πρώτο αντιπρόεδρο. Τρει συνεδριάσει του Τριλόγου διεξήχθησαν μέχρι τώρα. Επετεύχθη ουσιαστική πρόοδο σε πολλά πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε και θα τα περιγράψω συνοπτικά. Καταρχάς, όσον αφορά το μόνιμο σώμα, θέλουμε να φτάσουμε 10.000 προσωπικό επιχειρησιακό μέχρι το 2027. Πρόταση να δημιουργήσουμε και τέταρτη κατηγορία. Κάτι που έγινε καταρχήν ε, αποδεκτό. Παραμένουν οι αφορές στη δυνατότητα το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας δημιουργήσει μια ακαδημία εκπαιδευτική. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί ο μηχανισμός αναθεώρησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τα κάτι μέλη και το Συμβούλιο αυτό. Συμφωνήσω παραμείνουν οι διαγραφέ όλων των αναφορών στα κέντρα ελέγχου, διότι δεν έχουμε ακόμα ορισμό του σημείου αυτού. Καταφέρουμε να ισχύσουμε το ρόλο του υπευθύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διαθέτω κατάλληλου πόρου στον αξιωματούχο, να χρησιμοποιήσουμε και να έχουμε και έναν υπαξιωματικό ε, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπάρχει αυτονομία στο ρόλο αυτό το Συμβούλιο δέχτηκε την πρότασή μας να δώσουμε νέο ρόλο στα προσωπικά, στο προσωπικό της υπηρεσίας που παρακολουθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις ε, ε, εργασίες που εκτελεί η υπηρεσία. Θέλουμε το Συμβούλιο να δώσει επαρκή στελέχωση για αυτό το νέο ρόλο που θα παίξει η υπηρεσία, να ενισχύσουμε και τη δυνατότητα καταγγελιών σύμφωνα με θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρεται στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλία που ετοιμάσαμε η Σκά Κέλλερ και εγώ για τα διάφορα ε, διάφορα γραφεία σε τρίτες χώρες να δημιουργήσουμε τέτοια γραφεία και θα, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες επιχειρησιακές υπηρεσίες. Θέλουμε να κρατήσουμε τον παρόντα κανονισμό και το κείμενά του για τις ε, ομάδες υποστήριξης εφαρμογή του κανονισμού. Άλλο θέμα είναι η αναφορά στη δυνατότητα υπηρεσία να εμπλέκεται σε επιστροφές από μια τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα. Επιμένουμε επίσης ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται εμπλοκή ε, της υπηρεσίας λόγω κινδύνων θεμελιών δικαιωμάτων για δεύτερης απομακρύνσεις. Ελήφθη υπόψη πλήρωση η υπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφέρεται ότι η υπηρεσία δεν χρησιμοποιεί πόρους ούτω ώστε να υποστηρίξει η αδίποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με προσωπική ε, επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Τώρα, όσον αφορά τις διαδρομές, τους όγκους και περιορισμό διάδοση πληροφοριών, όταν είναι διαθέσιμο στις πληροφορίες στα κράτη-μέλη και αυτό έγινε δεκτό. Πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα, κυρίως για τη διακυβέρνηση και τη δίκηση αλλά πιστεύω ότι στους τριμερείς διαλόγους ε, θα πετύχω κάποια συμφωνία και ελπίζω να πιστέψει, η, η φωνή μου συγγνώμη τότε. Πάψτε να μιμήσετε την Πρωθυπουργό της Βρετανίας παρακαλώ. Ακούγεστε σαν Τερέζα Μέη, λέει και ο Στίμερμανς. Λοιπόν, δεν ήθελα να το πω αυτό τώρα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση Ρομπέρτα. Η Νάτα Ελίνη και η τη. Αν δεν θέλει να μιλήσει. Ο Πίτερ μετά. Ε, Πίτερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έγινε πολλέ συζητήσει συνεδριάσει των σχεδόν. Πολύ επικοδομητική η συνεργασία μας μεταξύ ε, του εισηγητή και της ομάδας μου. Εμείς υποστηρίζουμε απολύτως τη γραμμή του εισηγητή και λυπούμαστε που ενώ έχουμε πολύ καλές εξελίξεις επί το Frontex δεν γίνεται τίποτα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου ενώ αυτοί οι δύο φάκελοι είναι αλληλένδετοι. Δυστυχώ όμως δεν φαίνεται να υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση στο Συμβούλιο για να συζητηθεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Πάντως ε, ε, συμφωνούμε απόλυτα με τον εισηγητή και ελπίζουμε να βρεθεί μια καλή λύση τελικά ε, στις διαπραγματεύσει αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πίτερ και η εισηγήτρια που ήταν σχεδόν εισηγητής από το S&D έτσι. Και τώρα από την άλλη η κυρία Γκρίσμπεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλωσορίζω και τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς. Δύο λόγια και από την πλευρά μου σχεδόν εισηγήτρια να ευχαριστώ τη Ρομπέρτα που ακόμα και χωρίς φωνή ε, έχει κάνει πολλή δουλειά και έχει διαθέσει και πολλή ενέργεια ε, στον φάκελο αυτόν σε ένα πνεύμα συνεργασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε στην ε, ερχόμενη εβδομάδα να φτάσουμε σε μια συμφωνία που να ανταποκρίνεται στη βούληση μιας ευρείας πλειοψηφίας. Για τη δική μου πολιτική ομάδα αυτό μπορώ να πω είναι ότι παρακολουθούμε στενά ό,τι έχει να κάνει με την κατάρτιση. Ε, είμαστε κοντά στις σωστές διατυπώσεις νομίζω, αλλά και σε ό,τι αφορά την, το θέμα της σύνθεσης του Διευθυντικού Συμβουλίου. Αυτό είναι κάτι που θα καταστήσει την Frontex ε, μια υπηρεσία ε, πολύ σημαντική, την πιο σημαντική της Ένωσης. Θα βελτιωθεί και ο ρόλος της και η εντολή της και οι δυνατότητές της βέβαια. Συμφωνούμε λοιπόν απόλυτα με την εισηγήτρια και με τους και εισηγητές από αυτού. Υπάρχει ένα πολιτικό σημείο πολύ σημαντικό, το ρόλο, ο ρόλος της Frontex στην οργάνωση ε, της επιστροφής από τρίτες χώρες σε τρίτες χώρες. Είναι κάτι που είχε συζητηθεί και στην αρχή των εργασιών μας. Δεν ξέρω αν πρέπει να επιμείνουμε εδώ επ' αυτού, δεν είμαστε και πολλοί σήμερα εδώ. Να επενθυμίσω πάντως ότι ήταν σαφέστατη η θέση του Κοινοβουλίου και τη ομάδα μου τότε. Θεωρούμε ότι η υπηρεσία αυτή δεν ε, είναι ρόλος της να οργανώσει επιχειρήσει επιστροφής από τρίτη χώρα σε τρίτη χώρα. Δεν είναι δικό της ρόλος. Θα θέλαμε να επικεντρωθεί ε, στην δουλειά που πρέπει να γίνει στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ε, με δύο λόγια να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Ρομπέρτα, συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να φτάσουμε στη συμφωνία που ελπίζω να επιτευχθεί την ερχόμενη εβδομάδα όταν θα μπορέσουμε ε, να επιλύσουμε τα πολιτικά ζητήματα που εκκρεμούν έτσι ώστε ο κανονισμός αυτός να είναι παραδειγματικός, να είναι ένας πολύ ισχυρός κανονισμός. Ε, ευχαριστώ Νατάλη, ευχαριστώ και σένα Ρομπέρτα. Πριν περάσουμε στο σημείο της Ουγγαρίας, υπάρχει ακόμα ένα σημείο. Α, όχι, δεν θα το δούμε αυτό. Μάλιστα, εντάξει. Ε, φαντάζομαι ότι θα ανακουφιστεί και ο αντιπρόεδρο. Θα περάσουμε απευθεία λοιπόν στο θέμα 21, ε, στο σημείο 21 που αφορά την Ουγγαρία. Να καλωσορίσω για άλλη μια φορά τον αντιπρόεδρο Τίμερμαντ. Ε, συνάδελφοι, όπω γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο ανέκρινε μια, ένα ψήφισμα στις 12 Σεπτεμβρίου σε ό,τι αφορά την πρόταση προς το Συμβούλιο για το κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 7 της συνθήκης ε, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει σαφής κίνδυνος παραβίασης των αξιών πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση από την Ουγγαρία. Ε, αυτό είναι μια ευκαιρία σύμφωνα με την Επιτροπή Ελευθεριών τουλάχιστον να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις μετά την πρόταση ε, του Κοινοβουλίου. Συμμετέχει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είναι και ο κύριος Κάλιν Στάικα από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρουμανικής ε, Προεδρίας ε, και είναι και η Τζούντι Σαρτζεντίνη εδώ, η συγγήτριά μας και ε, οι συνεισηγητές που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους λοιπούς διακεκριμένους προσκεκλημένους. Να ξεκινήσω με τον Αντιπρόεδρο. Κύριε Τίμερμαντς, έχετε το λόγο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ελευθεριών που έθεσε το θέμα αυτό στην σημερινή μέρη στα διάταξη. Την περασμένη φορά που είχα ε, την τιμή να ενημερώσω το Κοινοβούλιο για τις κατάσταση στην Ουγγαρία ήταν στις 30, ε, στις, στις Ιανουαρίου στην Ολομέλεια. Εμείς ε, συμμεριζόμαστε μεγάλο αριθμό των ανησυχιών που εκφράζει η τελευταία πρόταση του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα Φορά... αφορά θεμελιώδη δικαιώματα, την καταπολέμηση τη διαφθορά, ε, τη μεταχείριση των Ρωμά και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να σε ενημερώσω για, για τι πρόσφατε εξελίξει, μετά τον Ιανουάριο δηλαδή, ε, και στο Συμβούλιο. Δυστυχώ η κατάσταση δεν βελτιώθηκε. Οι ανησυχίε που είχαν εκφραστεί στο παρελθόν δεν αντιμετωπίστηκαν και έχουν προκύψει και νέοι λόγοι ανησυχία έκτοτε. Προφανώ θα γνωρίζετε ότι το Φεβρουάριο η κυβέρνηση τη Ουγγαρία ξεκίνησε μια καμπάνια με μεγάλες αφήσει, διαφημίσεις σε εφημερίδες αλλά και επιστολή ε, του Πρωθυπουργού προς όλους τους Ούγγρους πολίτες με στόχο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον πρόεδρό της ε, τον κύριο Γιούνκερ. Αυτή η καμπάνια συνεχίστηκε παρά την ε, τις επικρίσεις που έλαβε από πολλές πλευρές η Κομισιόν ήταν σαφέστατη σε ό,τι αφορά αυτήν την άποψη στρεβλώνει την πραγματικότητα προσπαθεί να ε, να δώσει μια λαθασμένη και ε, μαύρη εικόνα της Ένωσης ότι υπάρχει δηλαδή μια συνωμοσία για να έρθουν περισσότεροι μετανάστες στην ε, Ουγγαρία. Εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε με την ίδια ισχύ όταν ακούγονται ψέματα, όταν η ρητορική που ακολουθείται είναι ψευδής και αυτό βεβαίως πλήττει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία απολύτως συνωμοσία. Νομίζω ότι οι Ούγγροι πολίτε δικαιούνται να μάθουν την αλήθεια, τα πραγματικά γεγονότα, σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών που είναι ο ιστό μιας δημοκρατικής κοινωνία. Είναι λοιπόν θεμελιώδες στοιχείο οποιοδήποτε κράτου μέλου της Ένωσης. Λυπάμαι που λέω ότι ούτε εκεί υπάρχει κάποια βελτίωση, σε καμία περίπτωση. Ε, μια ολόκληρη πανοπλία μέτρων έχουν πάρθει από τις αρχές και αφήνουν όλο και λιγότερο χώρο σε αυτές οργανώσεις. Τον Ιανουάριο αποφάσισε η Κομισιόν να στείλει μια γνωμο, γνωμοδότηση ό,τι αφορά την νομοθεσία στο ψώρος που ποινικοποιεί δραστηριότητε που βοηθούν τους ετούντε άσυλο ε, να θέσουν, να επιβάλλουν την υποψηφιότητά τους έως 24 Μαρτίου θα πρέπει να απαντήσει τι ανησυχίες της Κομισιόν η Ουγγρική Κυβέρνηση. η Κομισιόν ενδεχομένω να στείλει την υπόθεση αυτή στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, Στι 13 Φεβρουαρίου, πάντω, το Ευρωπαϊκό το, ε, Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων ζήτησε ε, να δοθούν τρόφιμα από τις Ουγγρικές αρχές σε δύο Ιρακινούς ε, οι οποίοι ήταν σε τράνζιτ στην Ουγγαρία ε, και που δεν έχει γίνει δεκτή η αίτηση ασύλου του. Δηλαδή να πρέπει να παρέμβει το, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να μπορέσουν να τραφούν δύο άνθρωποι στην Ουγγαρία. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα και βεβαίω φανταστείτε και τη δουλειά, τη σημασία της δουλειά, μιας ΜΚΟ που βοήθησε τους ε, άσυλο ε, στην περίπτωση αυτή. Τι θα είχε γίνει δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτή η ΜΚΟ. Ε, αναφερθήκαμε επίση. Ε, και στην ανησυχητική εξέλιξη όπου 400 διαφορετικά μίντια έχουν συγχωνευτεί σε ένα ε, και ελέγχεται από κάποιους διοκτήτες που είναι πολύ κοντά στο κυβερνόν κόμμα έγινε αποδεκτή η συγχώνευση ε, και δεν πέρασε ούτε από, η συγχώνευση αυτή ούτε από τον έλεγχο της αρχής ε, ανταγωνισμού ούτε από την αρχή ε, το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι πολύ ανησυχητική αυτή η κατάσταση. Δημιουργείται εδώ ένα νέο μηντιακό κατεστημένο. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε βεβαίω αυτή την κατάσταση και θα σα ενημερώνουμε σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση σε ό,τι την, του Πανεπιστημίου Κεντρική και Ευρώπη. Ούτε εδώ έχουμε θετικά νέα. Όπω είπα ήδη τον Ιανουάριο, ε, θα πρέπει το ακαδημαϊκό τη πρόγραμμα το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τι ΗΠΑ θα πρέπει λοιπόν να μετακομίσει στη Βουδαπέστη ήδη από το, από το 2019. Θα πρέπει να μετακομίσει από τη Βουδαπέστη στη Βιέννη. Το να υποχρεώσει κάποιο, ένα πανεπιστήμιο, να μετακομίσει τα προγράμματά τη ε, μετά από πιέσει μια κυβέρνηση είναι κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το ότι συνέβη κάτι τέτοιο παρά την διαδικασία που παραβάσει ε, που έχει ανοίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκρεμεί ακόμα αυτή η διαδικασία. Ε, σε ό,τι ε, αφορά την νομοθεσία για τις υπερορίες, την νομοθεσία της σκλαβιάς όπως ονομάζεται και με μεγάλες διαδηλώσεις, η, η, Ουγγρική κυβέρνηση έδωσε κάποιες διευκρινήσεις μετά από έτοιμά μα και εξετάζεται κατά πόσο πλέον μετά τι διευκρινήσεις αυτές η νομοθεσία συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Περιεργασία. Ό,τι διαφθορά, διαφθορά εξετάζουμε ε, την εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα που σχετίζονται με την ανάγκη να ενισχυθεί ε, το πλαίσιο τη διαφθορά. Η, έκθεση αναχώρα για την Ουγγαρία τη 20 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτω πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα του 2018 σε ό,τι αφορά την ανάγκη ενίσχυση του, του, του πλαισίου κατά της διαφθοράς, την αύξηση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στις δημόσιες προμήθειες. Επίσης, ε, τονίζουμε ότι με τις τελευταίες εξελίξεις υπάρχουν ανησυχίες ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια αξιολόγηση του δικαστικού σύστηματος της ε, Ουγγαρίας και λέγεται στην ανάλυση αυτή, στην αξιολόγηση, ότι υπάρχουν όλο και λιγότερα αντίβαρα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, ανεξαρτησία του Γενικού Εισαγγελέα θέλουμε να δημιουργηθεί ένα νέο ε, δικαστικό διοικητικό σύστημα στην Ουγγαρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Η Επιτροπή της Βενετίας συμφωνεί στην δική της νομοδότηση, θεωρεί ότι πολύ σημαντικές εξουσίες είναι στα χέρια λίγων εμπλεκομένων και δεν υπάρχουν αρκετά αντίβαρα ε, απέναντι σε αυτές τις εξουσίες. Ζητείται λοιπόν από την Ουγγρική Κυβέρνηση να τροποποιήσει την νομοθεσία της. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι με βάση την κριτική της ε, Επιτροπής της Βενετίας έχουν υποβληθεί ε, ήδη τροποποιήσει την περασμένη εβδομάδα στην νομοθεσία αυτή στον Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Ζητούμε από τι Ουγγρικέ Αρχέ να τροποποιήσουν την νομοθεσία για να καλυφθούν όλε οι συστάσει τη ε, Επιτροπή τη Βενετία. Θα παρακολουθούμε πολύ στενά τι νομοθετικέ αυτέ εξελίξει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα, ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνοντα υπόψη και την τη Επιτροπή τη Βενετία. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα τώρα για τη διαδικασία του άρθρου Βεβαίω το Συμβούλιο και η Προεδρία είναι αυτή που θα αποφασίσει πώ θα οργανώσει τι εργασίε τη. Λυπάμαι που έω τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δεν είχε την ευκαιρία να υποβάλει την πρότασή τη στο, Συμβούλιο, πρόταση στο Συμβούλιο. Η Κομισιόν έχει καταστήσει σαφέ ότι όποια και είναι η θέση του Συμβουλίου πρέπει να εξασφαλίσει μια ε, δίκαιη εξέταση ε, της πρότασης του Κοινοβουλίου. Ξέρετε, ε, ότι έχουμε παρουσιάσει και μια αξιολόγηση των γεγονότων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία παραβάση, το άσυλο, και και πολιτών, η ανώτατη εκπαίδευση και η ε, διακρίση στα σχολεία κατά τον Ρωμά. Υπάρχουν όλε αυτέ οι υποθέσει εκκρεμούν στο δικαστήριο. Για την ώρα η Ουγγρική κυβέρνηση έχει απαντήσει. Ε, δεν έχει απαντήσει μάλλον ακόμα σε αυτά τα ερωτήματα. Έχει όλα τα, τα, τα στοιχεία στα χέρια, της, στα χέρια του Συμβούλου να αρχίσει να αξιολογεί τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό και αναμένω το Συμβούλιο να επανέλθει στο θέμα αυτό στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ που αναφερθήκατε και στις εξουσίες του Κοινοβουλίου εν προκειμένου και δώσατε περισσότερη έμφαση σε αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε σε συνεργασία με το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Τώρα έχουμε τον κύριο Στόιτσα της ε, Ρουμανικής Προεδρίας. Ορίστε κύριε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Συμφωνούμε όλοι και θεωρώ την αυτονόητο και για την Ρωμανική Προεδρία ότι η προστασία του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της Ευρωπαϊκής μας Ένωσης Υπενθυμίζω στις 18 του πέρσι το Συμβούλιο δέχθηκε την αιτιολογημένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούσε από το Συμβούλιο να αναγνωρίσει τον σοβαρό κίνδυνο σοβαρής παραβίασης από πλευράς Ουγγρικής Δημοκρατίας των αξιών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτοτε το θέμα έχει επανέλθει δύο φορές μέσα στο 2018 στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και αρχές του φετινού χρόνου συζητήθηκε τον Φεβρουάριο ε, υπό Ρουμανική Προεδρία. Στις 12 Νοεμβρίου 2018, συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, λάβαμε από την Ουγγαρία την γραπτή της απάντηση στην αιτιολογημένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και μία της πράγμαση συμβα... Ε, ε, παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άνοιγμα διαδικασίας κατά της Ουγγαρίας. Σεπτέμβριο, τον Φεβρουάριο μάλλον φέτος, οι Υπουργοί συζήτησαν τα επόμενα βήματα που θα κάνουν στο θέμα αυτό και η επόμενη συνάντηση θα είναι στις 9 Απριλίου, όπως τόνισε προηγουμένως και ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε την αιτιολογημένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ να προκαταλάβω ούτε να εξάγω συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την τελική έκβαση της διαδικασίας. Ασφαλώς όμως θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. Και για το λόγο αυτό ο υπουργό μας ε, ευρωπαϊκών Υποθέσεων κύριο Τσάμπα συμφώνησε τον Φεβρουάριο να ενημερώσει εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα περιθώρια της επικείμενης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Στόιτσα για να μιλούμε ξεκάθαρα τώρα. Πρόκειται για ενημέρωση του Κοινοβουλίου, όπως είπατε, αλλά όχι για πρόσκληση του Κοινοβουλίου να συμμετάσχει στις συζητήσεις. Μα σα χρειάζεται μετάφραση. Λέει ο πρόεδρο. Αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έννοια ότι θα ενημερωθούμε. Εδώ όμω έχουμε συγκεκριμένε ρητέ εξουσίες και αναμένουμε πρόσκληση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα τονίσει και περαιτέρω η συγγετρία. Αλλά ήθελα να ακούσω από τα χείλη σας το τι δύναται να αναμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία βεβαίως βρίσκεται εν εξελίξη. Η εισηγήτρια θα, θα, θα εξηγήσει τα περαιτέρω. Θα ακούσαμε την εισηγήτρια και μετά συντονιστές και σκιώδεις. Όλα τα ονόματα αυτά είναι και γραμμένα στον κατάλογο. Θα, θα αρχίσουμε με την Τζούντι Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάντοτε είναι ευχαριστώ να ακούμε ότι θα ενημερωθούμε σε μια ε, ιστερότερη φάση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κύριο Τίμερμαν για την πλήρη επισκόπηση των όσων έχουν συμβεί το τελευταίο εξάμεινο λίγο πολύ. Έτσι ε, δεν είμαι αναγκασμένο να κάνω και εγώ το ίδιο. Όμως έχουν περάσει 6 μήνες μετά από την ψήφιση στις 12 Σεπτεμβρίου του ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εμεί ζητήσαμε τη σημερινή συνάντηση για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε. να κάνουμε ένα είδο απογραφή, το οποίο κάνατε. Όμως ιδίω προσκαλέσαμε ρητά την Ρουμανική Προεδρία για να μας εξηγήσει το χρονοδιαγραμμά της. Και πάλι τέτοιο πράγμα εγώ δεν άκουσα. Και δηλώνω την έκπληξή μου. Είχαμε τη Ρουμανική Προεδρία που ήλθε εδώ για να αυτοπαρουσιαστεί με δύο υπουργού ε, δικαιοσύνη και εσωτερικών. Και εγώ τους ρώτησα δημοσία, μπορείτε να μας διαφωτίσετε. Κάναμε και συζήτηση στην Ολομέλεια με συμμετοχή του Υπουργού του των Εξωτερικών. Πάλι τον, ή τον ρώτησα, μπορείτε να μα πείτε τι θα κάνουμε. Πήγα μετά και βρήκα την ίδια την Υπουργό και ρώτησα. Έχω έρθει και σε επαφή με την Ορμανική Πρεσβεία και ζήτησα συνάντηση που δεν δέχθηκαν. Και μόνο μετά από πολύ επιμονή δική μας μας επέτρεψαν μισή ώρα στον κύριο Μωράες και σε μένα πριν από τη συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και αρχικά μάλιστα μόνο τον κύριο Ρωμαία, ε, Μωράης δεν με είχαν δεχθεί να προσκαλέσουν και εμένα ως εισηγήτρια και ευχαριστώ τη γραμματεία για την επιμονή της και μέσα σε μισή ώρα υποτίθεται ότι θα λαμβάναμε μια ιδέα για το τι πρόκειται να κάνει η Ρουμανική Προεδρία. Όμως η Ρουμανική Προεδρία αντέστρεψε τα πράγματα και μας ζήτησε εμάς να τους ενημερώσουμε για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Μα έχουμε γράψει έκθεση και εσείς τώρα πρέπει να προχωρήσετε στη σχετική διερεύνηση. Είδα και χθε την συζήτηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι και αυτοί θα προχωρήσουν σε διερεύνηση με τρεις σοφούς ανθρώπους για να δουν τι γίνεται ακριβώς στην Ουγγαρία. Εμείς έχουμε κάνει τη σχετική δουλειά όμως και το επόμενο βήμα θα είναι να συζητηθεί σε βάθος στο Συμβούλιο. Ο πρόεδρος μας μίλησε ήδη για τα πράγματα αυτά, όμως το Κοινοβούλιο με επιστολή του ίδιου του Προέδρου του Ταγιάννη έχει ζητήσει και κατά επανάληψη μάλιστα να, κατα... να καταθέσουμε την έκθεση. Αυτό δεν έχει γίνει. Παραμένει ανοιχτό το θέμα αυτό. Αλλά, και θα το ξαναπώ, το Κοινοβούλιο δεν επιμένει να είναι παρόν σε κάθε συνάντηση του Συμβουλίου Υπουργών, παρόλο που εμεί έχουμε ανοιχτέ δημόσιε συζητήσει και εσεί είστε πάντοτε παρόντε εδώ. Δεν ζητούμε λοιπόν αυτό. Ζητούμε να βοηθήσετε στην αρχή τη διαδικασία σα. Διότι ναι, μεν ελάβατε την έκθεσή μα ήδη το Σεπτέμβριο, και όμω εξακολουθείτε να βρίσκεστε στην αρχή τη διαδικασία. Τη δική σα διαδικασία. Τον Φεβρουάριο μα είπε το Συμβούλιο ότι υπάρχουν ορισμένε χώρε μέλη οι οποίε δεν έχουν τόσο μεγάλη διάθεση να συζητήσουν το θέμα. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Δική σα όμω ευθύνη είναι να θέσετε το θέμα στην ημερησία διάταξη και να βάλετε και ένα χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να αφαιρεθεί θέμα από την ημερησία διάταξη παρά να εγγραφεί σε αυτήν. Η ερώτησή μου λοιπόν προ τη ρουμανική πρεσβεία, λέει η κυρία Σαντζετίνη, είναι γιατί δεν βάλατε χρονοδιάγραμμα, ποια βήματα θα κάνετε και πότε η πρώτη φορά που έθεσα την ερώτηση αυτή, η απάντηση που άκουσα ήταν ότι, ε, κοιτάξτε, μόλις άρχισε η Προεδρία μας και είναι πάρα πολύ ε, απασχολημένη. Τώρα όμως είμαστε στα μέσα της Προεδρίας σα σχεδόν, είμαστε το Μάρτιο και σας άκουσα προσεκτικά και δεν άκουσα απολύτω τίποτε. Και στο μεταξύ το θέμα αυτό μιλώ για ανθρώπους που δεν τους διατρέχουν, δεν τους διαθέτουν διατροφή και ενώ οι άνθρωποι κρατούνται. Οχτώ φορέ εκλήθη το δικαστήριο να κρίνει. Και μιλώ μόνο για τι υποθέσει που ξέρουμε. Η ΔΕ Επιτροπή Βενετία την προηγούμενη εβδομάδα μόλι κατέθεσε την ανάλυσή τη για τα νέα διοικητικά δικαστήρια στην Ουγγρική Δημοκρατία. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να αρχίσετε να κάνετε επιτέλου τη δουλειά σα και να δείτε τα νέα στοιχεία τα οποία εγώ δεν μπόρεσα να ε, ερευνήσω διότι η δική μου δουλειά τέλειωσε στις ε, 11 Σεπτεμβρίου και να τα περιλάβετε στις συζητήσεις σας. Αναμένω από εσά, κύριε Πρέσβη, να πείτε ποια είναι τα σχέδια της Ρωμανικής Προεδρίας και πώς προτίθεστε να διαρθρώσετε την συζήτηση. Τι είδους ενημέρωση να μου κάνετε, αν δεν μπορείτε να μου διευκρινίσετε από τα πριν, ποια είναι τα σχέδιά σας. Ιδού το βήμα που σας διαθέτουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ευρωβουλευτές που βρίσκονται εδώ για να πράξουν το δημοκρατικό καθήκον του που έχουν ψηφίσει και που έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους σε εσά. Με δύο τρίτα πλειοψηφία ψήφισαν οι ευρωβουλευτέ υπέρ του ψηφίσματος. Κύριε Πρέσβη, πέστε μας τι θα κάνετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαργεντίνη. πριν τον Αντιπρόεδρο και την Προεδρία, πριν δευτερολογήσουν, θα ακούσουν συντονιστές και τους και ηγητές. Η κυρία Σίπελ για τους σοσιαλιστές πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά σήμερα. Πριν να πω κάτι για την Ουγγαρία πιο συγκεκριμένα, θέλω να καταστήσω σαφές το εξή. Η Ουγγαρία είναι μια θαυμάσια χώρα η οποία αξίζει πάντοτε να την επισκεφθεί κανείς. Σε διάφορες ε, επισκέψεις μου στην Ουγγαρία γνώρισα εκεί πραγματικά καταπληκτικούς ανθρώπους και είναι σημαντικό να το πω αυτό ως εισαγωγή. Όμως αυτά που βλέπουμε εδώ και μία δεκαετία στην Ουγγαρία και όπου εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω κουραστεί να μιλώ για τα ίδια και τα ίδια. Και αυτό είναι κίνδυνος, διότι η κόπωση αυτή σημαίνει εν τέλει ότι κάπου συνηθίζουμε στις καταστάσεις αυτές. Και βλέπουμε παρόμοιες εξελίξεις και σε άλλες χώρες. Μιλώ για εξελίξεις για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ανεξαρτησία των μέσων επικοινωνίας, ανεξαρτησία της κοινωνίας των πολιτών. Ποινικοποιούνται οι προσπάθειες ανθρώπων που βοηθούν τους άστεγους, για παράδειγμα, τους πρόσφυγες. Και αφενός επί χρόνια δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα μετά ξεκινούν διαδικασίες επί παραβάση. Και ναι μεν ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όψη τεχνική να μην έχει άλλες δυνατότητες, αλλά τι θα πει infringement procedures ή αποφάσεις δικαστηρίων. Εν αμφιβολία ναι, κάποια στιγμή θα αλλάξει νομοθεσία. Όμως συχνά, σε πολλές περιπτώσεις, η ζημιά έχει διγίνει. Όπως για παράδειγμα η ζημια εχει γινει οπως για συνταξιοδότησης των δικαστών. Πράγματα που τα βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που βλέπω να λείπει από την δράση της Κομισιόν και βεβαίως ιδίω από το Συμβούλιο είναι μια ξεκάθαρη δήλωση διότι αυτά που κάνουν ο Όρμπαν και το κόμμα του είναι σαφέστατα και μονοσήμαντα όχι όπως λένε ορισμένοι πολιτικοί απλά ένα αστικό συντηρητικό κόμμα είναι αντιδημοκρατικό η συμπεριφορά αυτή είναι αντιδημοκρατική από την αρχή μέχρι του τέλους ξεκινούν με διέγερση παθών, ώστε μετά να εμφανιστεί ο Όρμπαν, ο αρχηγός τους, ως ο ισχυρός άνδρας που τα λύνει όλα. Και όταν εγώ επικρίνω το Συμβούλιο ότι απλώ κάθεται απαθής θεατής εδώ και χρόνια και δεν πράττει τίποτε, δεν ασχεί κριτική και θα το πω και καθαρά. Όταν προ 9 ετών, προ 8 ετών, ενδεχομένως και μάλιστα και πριν από 7 έτη, αν είχαμε τότε μιλήσει με καθαρή γλώσσα, θα υπήρχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κινηθούν οι εξελίξεις προς άλλη κατεύθυνση. Η σιωπή δεν αποτελεί πολιτική επιλογή. Και θέλω στη σημερινή συνάντηση, κανείς βέβαια δεν μπορούσε να τα προβλέψει από πριν, ότι θα υπάρξει σύμπτωση αυτή. Θέλω να επικρίνω ορισμένες γελίες συμπεριφορές και κάποιων πολιτικών κομμάτων. Δέκα χρόνια συζητούμε για την Ουγγαρία και Έχουμε, δεν έχουμε ακούσει τίποτε μάλιστα από τις ε, διάφορες κοινοβουλευτικέ ομάδες. Τώρα υπήρξε εκστρατεία με πλακάτ, με πανό και τώρα ξαφνικά, επειδή εμφανίστηκε εκεί και η φωτογραφία του Αντιπρόεδρου της Επιτροπής, ξαφνικά αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να βγάλουν τον Όρμπαν από το Λαϊκό Κόμμα. Για μένα είναι απολύτως αδιάφορο εάν ο Όρμπαν και τα μέλη του Φιντές είναι σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Με ενδιαφέρει ποια υποστήριξη δίνουν όλοι αυτοί. Αυτό που αναμένω ωστόσο είναι μια ξεκάθαρη γραμμή του Συμβουλίου και της Επιτροπής αλλά και μια ξεκάθαρη γραμμή από όλους τους επικεφαλείς κοινοβουλευτικών ομάδων και ιδίως από εκείνους τους επικεφαλείς πολιτικών ομάδων οι οποίοι έχουν βλέψεις και σε υψηλότερα αξιώματα να βγουν και να μιλήσουν για αυτά που συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Η σιγή τους και το να κοιτούν απλώς αλλού δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί στους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ Μπίρκιτ. Η κυρία Νάταλη Γκρίσπακ για το Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που μόλις υπόθηκαν από την Μπίκετ Σίπελ και από τον εισηγητή. Ο Λουί Μισελ που είναι ο σκιώδης στην ομάδα μας δεν έχει στην ουσία παρά ένα πράγμα να υπογραμμίσει που συμφωνεί συνοπτικά με αυτά που είπαμε. Μετά από όλα αυτά που έγιναν, μετά από τόσο χρόνο, τώρα που η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο κομβικό σημείο το Συμβούλιο δι, παίρνει μια θέση, επεξεργάζεται το θέμα και υποστηρίζει τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των τεκτενωμένων. Αυτό πρέπει να γίνει. Είμαι σύντομη, αλλά συμφωνώ με τις εργασίες που έγιναν. Είναι προσδοκία όχι των μελών μόνο της Επιτροπής, αλλά είναι προσδοκίες των Ευρωπαίων ε, που θέλουν να παραμείνει η Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Ναταλή για την ΚΟΕ. Η Μαρίν Κριστίν Βερζιά είναι σκιώδης επίσης για το θέμα αυτό η Κριστίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς. Έχω το προνόμιο, αν μπορώ να το πω έτσι, να παρακολουθώ από το 2010 ε, το θέμα. Είμαι σκιώδης για την ομάδα μου το 2010. Ομολογώ, πώς να το πω. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι κάτι κάπως σουραλιστικό. Να ξεκινήσω συμφωνώντας με αυτό που είπε η Μπίρκετ Σίπελ. Θα πρέπει κάθε φορά να το θυμόμαστε αυτό. Αυτό που κάνουμε εδώ ε, που επιθυμίζουμε τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα, ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι που στέφεται κατά των Ούγγρων, του Ουγγρικού λαού, αλλά κατά μια κυβερνήσεω που υπονομεύει του κανόνε του κράτου δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα των μέσων ενημέρωση και σωστά. Να σα υπενθυμίσω ότι το πρώτο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την Ουγγαρία αφορούσε ακριβώ το θέμα των μέσων ενημέρωση είναι του Μαρτίου 2011. Μιλήσατε για το θέμα της δικαστικής ανεξαρτησίας. Είναι σε σημαντικό κομμάτι ε, τμήμα του ψηφίσματος για δικαστική μεταρρύθμιση του Ιουλίου του 2011. Μιλήσατε για την Επιτροπή της Βενετίας, για το, για το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Τα συμπεριλάβαμε αυτά και από αυτής της βάσης ψηφίστηκε η έκθεση του Ιουλίου 2013 η έκθεση του κυρίου Ταβάρες. Σήμερα που βρισκόμαστε. Έχουμε 2019 παραμονές των ευρωπαϊκών εκλογών και θα πω ότι αν τα μέτρα, τα δέοντα είχαν ληφθεί και οι διαδικασίες επί παραβάση είχαν δρομολογηθεί από το 2011 σίγουρα δεν θα είχαμε φτάσει εδώ ούτε στην Ουγγαρία ούτε σε αρκετέ άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλο και περισσότερο αμφισβητούνται και υπονομεύονται. Όταν βλέπω ότι το ΕΛΚ επιτέλου τολμάει να ζητήσει κάποια, επιβάλλει ένα μέτρο αναστολή κατά του κ. Ορμπάν και θα προβεί σε νέα έρευνα για να δει τι γίνεται όσον αφορά την κατάσταση στην Ουγγαρία, λέω στον εαυτό μου, μα ποιον κοροϊδεύουν και κοροϊδεύουν πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα όλους τους Ευρωπαίους εκλογείς. Για μένα το θέμα του κάτω δικαίου της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θέμα θεμελιώδες. Είναι η βάση, είναι αυτό που συνέχεια λέμε, είναι η βάση του ε, οικοδομήματος Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν θέλετε να αποδείξετε πραγματικά αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεύθυνο για αυτά τα θέματα και όχι μόνο υποψήφιο των σοσιαλιστών για τι επόμενε ευρωεκλογέ, ζητώ συγγνώμη, αλλά ενημερώστε μας για την κατάσταση και κάντε κάτι πραγματικό, πραγματικά διαβήματα που έγιναν να μας πείτε. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δε, θα χρειαζόσαστε ε, να το κάνετε αυτό αν δεν υπήρχε πρόβλημα. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρκετά λόγια. Θέλουμε πράξεις σχεδόν με 10 χρόνια μετά ελάχιστα προχωρήσαμε και το κράτο δικαίου, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μονίμω υποχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι στο ύψο των περιστάσεων αυτών που συμβαίνουν. Ο αντιπρόεδρος σίγουρα θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θέλει τώρα ή αργότερα. Αργότερα. Εντάξει. Έχουμε άλλους δύο μιλητές. Τον κύριο Καλό και τον κύριο Νίτερ Μιούλερ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει. Ε, κύριε Γκάλ, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η συντονίστρια, η κυρία Ματσόλα, μου έδωσε το δικαίωμα να εκφραστώ, να μιλήσω για αυτήν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ήθελα όμως να πω τώρα αυτό που ήθελα να πω πριν. Να πω στον κύριο Τίμερμανς ότι δεν έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένο ότι σήμερα δεν μιλάμε για ένα νέο ψήφισμα κατά της Ουγγαρίας. Εν τη την περιπτώση πρέπει να πω ότι έπρεπε, καθήκον του ήταν, να μας πει τι γίνεται στο Συμβούλιο όσον αφορά τη διαδικασία. Πιστεύω ότι Σήμερα πήρατε περισσότερο χρόνο, είχατε χρόνο στη διάθεσή σας. Και βλέπουμε ότι δεν ακολουθείτε μια αντικειμενική προσέγγιση στο θέμα. Πρόκειται περί πολιτικής συνωμοσίας εναντίον μας εκ μέρους της αριστεράς και εκ μέρους της κυρίας Αργεντίνη. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν αφορά το όλο ζήτημα μόνο την Ουγγαρία, διότι αναφερθήκατε και σε κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στο slave law, όπως αποκαλείται. Θα πρέπει να γνωρίζετε ονομόνο η Ουγγρική αντιπολίτευση αναφέρεται σε αυτό το νόμο, αποκαλώντας το νόμο της δουλείας, νόμο της κλαβιάς. Αυτό αποδεικνύει ότι εσείς μιλάτε στα πλαίσια προεκλογικής εκστρατείας και κατά την άποψή μου αυτό είναι αξιόμεμπτο. Να προσθέσω ότι όλα αυτά που εσείς είπατε κατά του κράτους δικαίου, για την κατάσταση την κακή για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, όπως διατείνεστε, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κάτι άλλο παρά για πληροφορίες που δόθηκαν από κάποιους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Εσείς αναφέρεστε σε αυτά τα γεγονότα, σε αυτά τα στοιχεία μόνο για να τονίσετε και να στηρίξετε τους στόχους σας, τους στόχους της προεκλογικής σας εκστρατείας. Εγώ δεν πιστεύω το πρόβλημα ενός πανεπιστημίου που μπορεί να δώσει αμερικανικό ή ουγγρικό ε, πτυχίο είναι ένα πρόβλημα που είναι ένα πρόβλημα κράτους δικαίου. Εγώ πιστεύω ότι αν η απόφαση να απόκειται στο Συμβούλιο ας αφήσουμε το Συμβούλιο να κάνει τη δουλειά του για να υπάρξει μια αντικειμενικότητα και να υπάρξει και ο σεβασμός από πλευράς των διαφόρων θεσμικών οργάνων, χωρίς να γίνεται μια προεκλογική εκστρατεία. Να επιστήσω την προσοχή σε επίσης ότι σήμερα δεν συζητούμε εκ νέου ένα πρόβλημα της Ουγγαρίας. Σήμερα δεν πρέπει να μιλάμε εκ νέου για την Ουγγαρία. Δεν πρόκειται περί τηλεοπτικής σειράς που όλοι πλέον ε, παρακολουθούν και έχουν κουραστεί. Όμως εσείς δυστυχώς αυτό δεν το σέβεστε. Είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου σε όλες τις συνεδριάσεις αυτής της Επιτροπής και στο Κοινοβούλιο όλες οι συνεδριάσεις να χειραγωγούνται από την κυρία Σαρτζεντίνη και από άλλους για να κάνουν μια πολιτική εκστρατεία, μια προεκλογική εκστρατεία. Κατά την άποψή μου όλα αυτά που υπόθηκαν εδώ έχουν ξεπεράσει τα όρια που είχαν αποφασίσει οι συντονιστές. Ευχαριστώ. Ναι, για να είμαστε σαφείς, ε, ο αντιπρόεδρος είναι εδώ κατόπιν ε, δικής μας ε, πρόσκλησης. Το άρθρο 7 έχει βεβαίω βεβαίως ε, ενεργοποιηθεί πολύ καιρό πριν από τα τελευταία γεγονότα και η κυρία Σταντιστίνη επίσης δεν είναι υποψήφια σε ευρωεκλογές. Ο κύριος Νίντερ Μιλλερ είναι ο τελευταίος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Τίμερμαντς είπε ότι το τελευταίο διάστημα η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα και ότι έχει επιδεινωθεί σε πολλές περιπτώσεις. Και έτσι είναι κατά κάποιο τρόπο. Η κυβέρνηση όλο και πιο επιθετικά παραβιάζει την νομιμότητα. Το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ούτε καν δέχεται να συζητήσει μια πρόταση της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μάλιστα επιβάλλει κυρώσεις ε, σε βουλευτές της αντιπολίτευσης. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ε, στην ενημέρωση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πανεπιστήμιο το οποίο κινδυνεύει. Γενικά η ακαδημαϊκή κοινότητα της Ουγγαρίας, όλο το ακαδημαϊκό δίκτυο ε, απειλείται. Ο τομέας της έρευνας επίσης δέχεται συνεχείς πιέσεις, εκβιασμούς. Η κυβέρνηση λέει στους ερευνητές πού πρέπει να κάνουν έρευνα. Ο τομέας ο ακαδημαϊκός, ο επιστημονικός της έρευνας στην Ουγγαρία δεν λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που συνέβησαν χθες στο ΕΛΚ. Είπαν οι επικεφαλής του ΕΛΚ ότι η πολιτική που εφαρμόζει το ΦΙΝΤΕΣ δεν συνάδει με τις αξίες του ΕΛΚ. Συντηρητικές αξίες, χριστιανικές αξίες. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι το ΦΙΝΤΕΣ δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι το κόμμα που κυβερνάει στην Ουγγαρία. Όταν λοιπόν το ΕΛΚ λέει ότι αυτή η πολιτική του ΦΙΝΤΕΣ δεν συνάδει με τις αξίες του, τις συντηρητικές και χριστιανικές, αυτό ισχύει και την Ουγγρική κυβέρνηση, το σύνολό της διότι είναι το ίδιο πράγμα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό μόνο. Μπορεί να φανείς ο κύριο Γιούνκερ, η κυρία Τίμερμαν, η κυρία Σαρτζεντίνη, στι αφήσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται με χρήματα από τους Ούγγρους πολίτες. Τι θα συμβεί με αυτή την τριμελή επιτροπή που δημιούργησε το ΕΛΚ, τι θα συμβεί τελικά με την Ουγγαρία, τι θα αποφασίσει για την Ουγγαρία, τι θα αποφανθεί και οι αποφάσεις που θα πάρει πώς σχετίζονται με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να περάσω τώρα στο, στο Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που έχουν λάβει η χώρα το τελευταίο διάστημα και που έχουν επηρεάσει ε, σημαντικά την Ευρώπη. Η προσφυγική κρίση και η παραβίαση του κράτους δικαίου. Σε ό,τι φορά τους πρόσφυγες, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να πάρει οποιαδήποτε απόφαση τους ήταν αδύνατο να φτάσουν σε συνένεση. Το Συμβούλιο λοιπόν δεν έκανε τίποτα αν κάτι επηρεάζει περισσότερο τη φήμη, την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακριβώς αυτή η απραξία του Συμβουλίου. Και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στη Ρουμανική Προεδρία, γιατί η Αυστριακή Προεδρία τι έκανε, απολύτως τίποτα. Δεν συζητούμε λοιπόν εδώ ένα απομονωμένο γεγονός το Συμβούλιο δεν έχει πολιτικό θάρρος, δεν καινοτομεί ποτέ στη λήψη αποφάσεων και αυτό βεβαίως πλήττει ε, γενικότερα την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, νομίζω όταν μιλάμε για δράση και για αδράνεια ε, είναι συχνά το Συμβούλιο αυτό που είναι κοντά στην Αδράνη. Το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα που προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να εκφράσω για πίεση προ την Προεδρία, απλώ ήθελα να το πω αυτό. Σα ευχαριστώ για τι συνεισφορέ σα. Θα το ζητήσω τώρα από τον κύριο Αντιπρόεδρο να απαντήσει και από την Προεδρία βέβαια και στο τέλος μπορεί να παρέμβει και η συγκέντρια εν συντομία. Παρακαλώ κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μπορεί να μην κατάλαβα εγώ καλά την πρόσκληση της ΛΥΜΠΕ. Νόμιζα ότι είχα προσκληθεί για να παρουσιάσω στη ΛΥΜΠΕ το πού βρισκόμαστε. Και έδωσα τις πληροφορίες που έχω εγώ για το τι έχει αλλάξει, τις εξελίξεις σε από την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο πριν από μερικούς μήνες. Και αυτό ακριβώς έκανα. Δεύτερον, ε, θα ήθελα να γνωρίζω, αφού του άκουσα την κυρία Γκάλ, εάν μιλάει στο όνομα του ΕΛΚ. Το σύνολο του ΕΛΚ, έτσι. Θα ήθελα πραγματικά να το ξέρω αυτό, θα το έχω κατά νου όταν θα έχουμε συζητήσει το κράτο δικαίου, αν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι μερικά τα πράγματα που η κυρία Γκάλ ε, δεν έχουν θέση σε, σε αυτά που λέει το ΕΛΚ ή κάποιοι άλλοι από το ΕΛΚ. Λέει ότι μιλάει στο όνομα τη ομάδα τη, Αν είναι έτσι, πραγματικά εγώ θα σημειώσω πολύ προσεκτικά όλα αυτά που είπατε και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά τους επόμενους μήνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι συνέβη πριν την ε, Επιτροπή Juncker, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, διότι το θέμα αυτό όντως μας απασχολεί εδώ και 10 χρόνια περίπου. Είναι δύσκολο όμως εγώ να αναλάβω την ευθύνη για πράγματα που έγιναν ή δεν έγιναν πριν αναλάβω τα καθήκοντά μου. Και θέλω να πω για την περίοδο που ήμουν εγώ υπεύθυνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κράτου Δικαίου, ε, ευσυνείδητα προσπάθησα να παρακολουθώ όλα όσα εμείς θεωρούμε ότι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις της Ουγγαρίας απέναντι στις συνθήκες. Το παρακολουθούμε με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όντω η διαδικασία επί παραβάση παίρνει χρόνο. Η διαδικασία επί παραβάση όμως είναι και ένα ισχυρό μέσο, διότι δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με το κράτος μέλος. Και αν ο διάλογος δεν οδηγήσει στα αποτελέσματα που προσδοκούμε, τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι αυτό που κρίνει κατά πόσο υπάρχει παράβαση της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ή όχι. Και σε σχέση με το θέμα της Ουγγαρίας, έχει αυτό πιάσει τόπο και έγιναν κάποιες διορθώσεις για κάποια σημεία που εμείς, όπου εμείς θεωρούσαμε ότι η Ουγγαρία δεν ευθυγραμμίζεται με τις υποχρεώσεις της, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να κάνω τώρα ένα σχόλιο για τις γενικότερες εξελίξεις, διότι ε, διαπιστώνω ε, ότι βεβαίως πρέπει να λέμε για κάποιες αλήθειες που πονάνε, ε, υπάρχει μεγάλη υποστήριξη στην Ουγγρική κοινωνία για τις δράσεις ε, της, Ουγγρικής, κυβέρνησης. Διότι η Ουγγρική κυβέρνηση με διάφορους τρόπους έχει καταφέρει ε, να αλυσοδέσει τους Ούγγρους τους φόβους τους. Το φόβο ιδιαίτερα των μεταναστών και των προσφύγων. Όμως σας παρακαλώ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείτε να λέτε ότι περασπίζετε τις χριστιανικές αξίες, το χριστιανισμό και την Ευρώπη και ταυτόχρονα να αρνείστε να δώσετε νερό και τρόφιμα σε ανθρώπους που έχετε υπό την επίβλεψή σας. Πώς συνάδουν αυτά τα πράγματα. Καλωσορίζω λοιπόν όσους είναι υπέρ χριστιανικών αξιών αλλά να γίνει και μια συζήτηση τελικά. Ποιε είναι αυτέ οι χριστιανικέ αξίε. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα την Πρόεδρε. Ο κύριος Στόικα μήπως θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς να υπενθυμίσω κάτι. Η Ρουμανική Προεδρία διεξήγηκε μια συνάντηση πριν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 19ης Φεβρουαρίου. Αντιλάγησαν πληροφορίες με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση όσον αφορά την πρόταση που υπευλήθη πρόσφατα στο Συμβούλιο. Το χρονοδιάγραμμα. Η Προεδρία πράγματι καθορίζει το πρόγραμμα σε στενή διαβούλευση όμως με όλα τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτό στη διαβουλευτική διαδικασία που την ακολουθήσαμε, καταλήξαμε ότι δεν θα πρέπει να εξαχθεί συζήτηση επ' αυτού του σημαντικού θέματος στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του Μαρτίου. Να επιβεβαιώσω εκ νέου ότι περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων προβλέπεται για το επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 9 Απριλίου, όπως ανέφερα προηγουμένως. Να μοιραστώ μαζί σας κάποιες τεχνικής φύσεως πτυχές όσον αφορά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία. Θα θυμόσαστε ίσως ότι το άρθρο 7.1 δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο βασικά προνόμια. Κανένα από αυτά προβλέπει συμμετοχή όμως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συζητήσεις του Συμβουλίου ούτε από πλευράς ε, βοηθείας ούτε να ε, γίνει μια προφορική παρουσίαση πρόσφατης προτάσεις. Όσον αφορά τη συμμετοχή στη συζητήση του Συμβουλίου, αυτό είναι κάτι που ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου. Και έχω εδώ ένα σημείωμα για το άρθρο 5.2 που αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φερρυπίν θα κληθεί να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ίδιο ισχύει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε περιπτώσεις όπου ασκεί το δικαίωμα αυτή, το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Καμία τέτοια πρόβλεψη δεν υπάρχει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν από το Κοινοβούλιο υπέβαλε κάποια πρόταση, το Κοινοβούλιο δεν προσεκλήθη να συμμετάσχει σε επίσημες συζητήσει του Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν εμπόδισε μια καρποφόρα συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, να πω ότι οι θεσμικές ρυθμίσεις όσον αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου που συνέταξε την πρόσφατη πρόταση και το προνόμιο να δώσει σύμφωνη γνώμη ε, επιτρέπει να έχει ένα σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο στη λήψη τελική απόφαση, όμω απαιτείται και συνεργασία με το Συμβούλιο. Κάτι που προσπαθεί να ακολουθήσει ενεργά η Προεδρία. Δεν υπάρχει δυστυχώς περιθώριο για άμεση συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε επίσημες συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Μακάρι να μην τα είχατε πει όλα αυτά. Τι θέλατε και τα είπατε αυτά δημοσία, κύριε Στόικα. Σοβαρά μιλάω τώρα. Δύο επιστολές. Πρέπει να ξέρετε, το συζητήσαμε λεπτομερό το θέμα. Αν θέλετε αυτό να συζητηθεί ανοιχτά στην Επιτροπή μου, με τα χαράς να το κάνω, και ενώπιον του πρώτου Αντιπροέδρου ζητάμε τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Ποια είναι τα, τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Είχαμε δύο ε, επιστολές που στείλαμε από τον Πρόεδρο. Τι λέτε δηλαδή. Ότι στον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου υπάρχουν και άλλοι κανόνες που λέει ότι οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο μπορεί να προσκληθεί. Αλλιώς τι γίνεται, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάει στο ΕΚΟΦΗΝ ή άλλες υπηρεσίες πάνε στις συνεδριές του Συμβουλίου κυρία Σαρτζεντίνη και εγώ να μην κολλήσουμε σε μια, κολλήσαμε, να κολλήσουμε σε μια αίθουσα, να μας τριμώξετε σε μια αίθουσα 9 Απριλίου. Ας μας καλέσετε τουλάχιστον μία φορά στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για να συνεχιστεί η δουλειά που κάποια μέλη, κάποια άλλοι συνάδελφοι ίσως θεωρούν ότι δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα. Και ίσως αν ε, μα επέκρινε ο πρώτο αντιπρόεδρο, δεν προχωράμε αρκετά γρήγορα. Κάνουμε εμεί τη δουλειά μα συνεργαζόμενοι για να προχωρήσουμε. Λυπούμε, θα μπορούσα να πω και περισσότερα και να βαρεθούν όλοι. Ίσως η κυρία Σαρτζεντίνη μπορεί να κάνει όλους να βαρεθούν. Αυτό όμως δεν ισχύει αυτό που είπατε. Πηγαίνετε, εξετάστε τις επιστολές που στείλαμε και είναι απαράδεκτο να βρισκόμαστε ε, σε αυτή τη θέση. Δεν πρέπει να ενημερωνόμαστε. Έχουμε επίσημο ρόλο σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία. Δεν πρόκειται περί απλή ενημέρωση. Με εκπλήσει που το λέτε αυτό ανοιχτά. Δεν ξέρω αν ο πρώτος αντιπρόεδρο έχει κάποια άποψη επ' αυτού. Ο κ. Τίμερμανς, δύο πράγματα να πω. Το πρώτο είναι γενικότερο. Όταν συντάχθηκε η συνθήκη και το άρθρο 7 και το άρθρο 50, ας προσθέσω αυτό, εγώ συμμετείχα στη διαδικασία, τότε κανεί δεν θεωρούσε ότι θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα άρθρα. Ξεπερνούσε ε, την πραγματικότητα της ε, φαντασίας ότι θα πρέπει να στραφούμε κατά ενός κράτους μέλους γιατί σέβεται το κράτος δικαίου, ότι κάποιο κράτος μέλος θέλει να αποχωρήσει. Όταν συνετάχθησαν δεν μπήκαμε σε επαρκές βάθος όσον αφορά την πλήρη ανάλυση των συνεπιών της πλήρους εφαρμογής του άρθρου. Τώρα για το άρθρο 7 δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εσωτερικό κανονισμό για να εμποδίσουμε ένα από τα θεσμικά όργανα να παίξει τον πλήρη ρόλο του, αν ο ρόλος αυτός αναφέρεται στο άρθρο 7. Αυτή είναι η γενική μου παρατήρηση. Πιο συγκεκριμένη παρατήρηση. Επειδή κάποιοι στο Συμβούλιο και κάποιοι, κάποια, νομική, κάποιοι σύμβουλοι στο Συμβούλιο επιμένουν ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επιτραπεί να το κάνει αυτό, μετά στρέφονται προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δώσει τι πληροφορίε ή να κάνει κάτι. Αυτό δεν το δέχομαι. Δεν θα με βάλετε στη θέση στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει τη δουλειά του Κοινοβουλίου. Ε, αυτό δεν είναι σεβασμό απέναντι στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο πήρε μια απόφαση για το άρθρο 7, κυρίαρχη απόφαση. Και το Κοινοβούλιο, κατά την άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει γιατί έχει αυτή τη θέση, να τονίσει τα διάφορα σημεία που επιθυμεί στο Συμβούλιο. Διότι τώρα το Συμβούλιο σε κάποια φάση θα πρέπει να λάβει μια απόφαση σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, δεν θέλω εγώ τώρα να παρασύρετε σε όλα αυτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι υπάρχει σαφήνεια μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σχετικά με το πώς μπορεί να εκπροσωπηθεί το Κοινοβούλιο Συμβούλιο. Ένα ε, γενικό σημείο και το δεύτερο πιο ειδικό που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είμαστε διαμεσολαβητή, δεν εκπροσωπούμε, δεν είμαστε φερέφωνο του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει δική του φωνή και δεν θα μας βάλετε, κανείς δεν θα μας βάλει σε αυτή τη θέση. Επίσης, να προσθέσω Είπατε ότι ήταν νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Το αμφισβητώ. Ήταν προφορική γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Δεν ήταν επίσημη γνωμοδότηση γραπτή του Συμβουλίου. Δικαιό. Σωστά. Έτσι. Δεν ήταν νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Η κυρία Σαρτζεντίνη σου τον έφερε πριν. Δεν λέμε ότι θέλουμε να εμφανιζόμαστε κάθε δύο λεπτά. Έτσι μας αντιμετωπίζουν. Μια φορά θα αρκούσε. Αλλά δεν θέλουμε να αντιμετωπιστούμε με δύο ενημερώσεις σε, μια, σε ένα δωματιάκι όπως είπε ο Αντιπρόεδρος να χρειαζόμαστε ε, διαμεσολαβητές. Είναι προνόμιό μας. Την επόμενη φορά όταν έρθετε παρακαλώ να έχετε επίγνωση ότι ξέρουμε τη συζήτηση και δεν μπορείτε να μας απορρίπτετε έτσι. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρε. Χαίρομαι πολύ για τα όσα είπατε και ευχαριστώ και εσάς κύριε Αντιπρόεδρε που μπαίνετε στον καυγά. Δεν υπάρχει ωστόσο νομική γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Ε, πρόκειται μόνο για μια προφορική τοποθέτηση. Και μέσω αιτήσεων από πολίτε για πρόσβαση σε έγγραφα, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει τέτοια νομική γνωμοδότηση. Τώρα, εγώ βλέπω και μία τάση μέσα από την έκθεσή μα. Ε, εξήγησα πια την μεθοδολογία εργασία μου με δήλωση ώστε κανείς να μην μπορεί να την αμφισβητήσει. Και επειδή πρέπει να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία και μέρος της διαδικασίας αυτής είναι να αποδεχθούν και στο Συμβούλιο ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας. Πρόκειται για διαδικασία του άρθρου 7. Δεν ε, ζητούμε απλά εμείς να είμαστε παρούσες και παρόντες σε κάθε συνεδρία του Συμβουλίου. Όχι, υπάρχει το άρθρο 7 και δεν προβλέπεται καμιά ιεραρχική ε, δεν υπάρχει καμιά ιεραρχική ε, κατάταξη των θεσμικών οργάνων για το ποιο θα αρχίσει την πρωτοβουλία. Αλλού άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί αρχίσαμε για την Ουγγαρία και εσεί θα μπορούσατε να είχατε αρχίσει και θα ήσασταν βέβαια και ταχύτεροι εσεί ω Συμβούλιο δηλαδή. Δεν υπάρχει λοιπόν ιεραρχική κατάταξη, ξαναλέω, στην συνθήκη για το ποιο θεσμικό όργανο ξεκινά την διαδικασία. Έχω την αίσθηση ότι το Συμβούλιο κάπου βλέπει μια τέτοια ιεραρχική κατάταξη που δεν βασίζεται στο γράμμα του άρθρου. Και είναι πολύ ενοχλητικό που το Συμβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέλθει, αλλά τη ζητεί και επισκόπηση, επισκόπηση των, των διαδικασιών έχει παραβιάση. Ενώ το Κοινοβούλιο βλέπει μια πολύ ευρύτερη οπτική, γιατί μιλούμε για τις βαριές επιπτώσεις στην κοινωνία όλων των πτυχών που έχουμε αρχίσει να συζητούμε ήδη από το 2010 και πράγματα που κάνει δηλαδή η Ουγγρική κυβέρνηση. Με ε, μιλείτε εσείς για γόνιμη συνεργασία και ενεργό προσέγγιση από πλευρά σας προς εμάς. Εγώ έχω άλλη έννοια για το τι σημαίνει καρποφόρα συνεργασία και proactive. Εμείς τίναμε χείρα συνεργασία σε τέσσερις υπουργούς. Εσείς Ούτε προακτιβήσασταν, ήσασταν, ούτε συνεργασία δείξατε. Αρνηθήκατε να με συναντήσετε. Ξαναλέω, θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα να μας προσκαλέσετε στις 9 Απριλίου να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχουμε κάνει. Αυτό είναι το ένα. Δεν θα το δεχτείτε κατά πάσα πιθανότητα. Το άλλο που θα θέλαμε είναι, θα θέλαμε και σας έχουμε δώσει ως τώρα πέντε ευκαιρίες δημοσία να μας εξηγήσετε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας. Δηλαδή πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε τα διαφορετικά θέματα που θέτει το άρθρο 7. Αρνηθήκατε να το πράξετε. Εγώ το βλέπω αυτό ως σημάδι μη διάθεσης προς συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα μας δεχτείτε με μεγάλη χαρά ως προσκεκλημένους. Αλλά θα δω ξανά τον Πρόεδρο γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για απαράδεκτη κατάσταση, ότι δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξουσίε του Κοινοβουλίου προ το τέλο τη κοινοβουλευτική θητεία. Και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο τη Κομισιόν που διευκρίνησε για άλλη μια φορά τι θέσει μα. Σα ευχαριστώ κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Επιθυμεί άλλο κανεί να τοποθετηθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώτο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίο προσεκλήθη. Ευχαριστώ και την Προεδρία. Αντιλαμβάνομαι ότι αντιμετωπίσατε περισσότερα από ό,τι αναμένατε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Θεμελιδών Ελευθεριών. Εδώ ε, λίγη συνεδρία. Ευχαριστώ.